προστασία της υγείας η οποία συνδέεται και με την προστασία των ζώων των όντων και θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία ε, Σάιφη για την εκθέση.